Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Λαμασούρ. Εφαρμογή των διατάξεων των συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία. Καταρχήν θα ψηφίσουμε την τροπολογία 2 της παράγραφου 9 με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Και πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάω στο δεύτερο τμήμα της παράφου 12 με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16 του αρχικού κειμένου. Μια ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19 του αρχικού κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20 του αρχικού κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 36. Τροπολογία 4 με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 36 με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, ξεκινάει η ονομαστική ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος Γ της ε, τελικής έκθεσης τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου κατά αποχές εγκρίνεται. Στο δεύτερο τμήμα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε στο σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχί, αρχίζει, τελειώνει. Εγκρίνεται. Και τώρα να δώσουμε σύντομα το λόγο στον συνάδελφο Λαμασούρ. Ε, συνάδελφε Λαμασούρ, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους σχεδόν τους συναδέλφους που υπεψήφισαν την έκθεση και κατ' εξαίρεση ζήτησα το λόγο, διότι είναι... Ε, Όλο τυχαίω, η τελευταία έκθεση την οποία ανέλαβα για την Ολομέλεια μετά από 27 χρόνια παρουσίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Αλλά θα σας βρω και μια τιμωρία. Με δύο επιπλέον στοιχεία. Το 1989 ήρθα εδώ σε ένα τότε πολιτικό φόρουμ που περιοριζόταν σε ένα μέρος της Ευρώπης δυτικά του σιδερένιου παραπετάσματος. Το κοινοβούλιο από το οποίο θα φύγω σε λίγες εβδομάδες είναι ένα πραγματικό κοινοβούλιο, ε, πλήρως ευρωπαϊκό, με νομοθετικές αρμοδιότητες. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ξεκινώντας από την ομάδα μου φυσικά, αλλά και πέραν της ομάδας μου, τους συνεργάτες του Κοινοβουλίου, των πολιτικών ομάδων, τους βοηθούς μας, για όλη τους την δουλειά για την κοινή μας δουλειά. Και χάρη σε εσά, συνάδελφοι, έμαθα, διδάχθηκα ότι τον ακούει κανείς, να οργανώνει διάλογο, να δείχνει ε, σεβασμό, να ψάχνει συμβαστικές λύσεις, ε, αιμονικά να ψάχνει το κοινό συμφέρον, είναι τα αποτελεσματικότερα μέτρα από ότι η συστηματική αντιπαράθεση που πολλές φορές είναι το ίδιο των εθνικών μας κοινοβουλίων. Πολύ, πολλά από τα εθνικά μας κοινοβούλια όπως και το εντυπωσιακό το ε, ε, Καπιτόλιο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα είχαν πολλά να μάθουν εδώ στο Κοινοβούλιο. Παραμένουμε προτεργάτες, ανώνυμοι, ταπεινοί αλλά υπερήφανοι ε, που προσφέραμε αυτό το λιθαράκι σε ένα πολιτικό οικοδόμημα που θα σημαδέψει την ιστορία της Επίρου μας. Στο μελλοντικό Κοινοβούλιο στο οποίο δεν θα έχω πλέον την τιμή να είμαι μέλο. Ελπίζω η πλειοψηφία που, ε, θα εκφραστεί, που εκφράστηκε τώρα θα είναι ενωμένη για να μπορέσει να προσαρμόσει την ενωσή μα στι προκλήσει του νέου αιώνα. Ευχαριστώ και πάλι. Έχετε την αμέριστη υποστήριξή μας σε όσα είπατε και για το μήνυμα που μεταφέρατε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας τριακονταετού δουλειάς, σε εσά τον ίδιο εκφρασμένο. Το σώμα σας εύχεται ε, κάθε τύχη στο μέλλον σας και στη ζωή σας. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Μπρέσο. Ε, εφαρμογή των διτάξεων των συνθήκων που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή. Ψηφίζουμε το παράγραφο 4, τροπολογία 2, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Παράγραφος 4. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 3. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 8, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10, τροπολογία 4, υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24. Αρχικό κείμενο ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 22, τροπολογία 6, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26, τροπολογία 5, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 28, αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 36, τροπολογία πρώτη. Ονομαστική εκκλησία άρχεται αυτή. Πέρας. Απορρίπτεται. Εταιρεολογική σκέψη D, αρχικό κείμενο, ονομαστική εκκλησία έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία Κ. Και αρχικό κείμενο. Γνωστή κλίση άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση της συναδέλφου Σπινέλη. Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωτών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο θεσμικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράγραφο 2, τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 2, τροπολογία 8. Ονομαστική κλίση. Άρχεται αυτή. Πέρα. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 8, τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ε, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 9, τροπολογία 5. Ονομαστική κλίση άρχεται αυτή. Πέρας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 9, τροπολογία 9, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 10. Επέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 14, παράγραφος 6, ονομαστική κλίση. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 17, τροπολογία 11, ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 21. Τροπολογία 7, ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 21, τροπολογία 12, ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 26, τροπολογία 13, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Επίση μετά την παράγραφο 26. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. 14 άρχεται πέρας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 27, πρώτη τροπολογία, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 28, 2, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 28, τροπολογία 15, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 15, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απολύτωται. Παράγραφος 32, τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 42 του αρχικού κειμένου ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση. Του κυρίου Ρανζέλ καθεστώ και γενική όρια άσκηση των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καθεστώ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Άρθρο 1, παράγραφος 3, τροπολογία 3, ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε τροπολογία 23 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Άρθρο 2, παράγραφος 7, τροπολογία 4, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Ας ελέγξουμε. 18. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Παρακαλώ. 19. Έλεγχος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 καταπίπτει. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Ακούω αυτή την πτέρυγα και μια χοροδία. Ας ελέγξουμε. 30. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν μπορώ να πω και να αποφασίσω. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 3, παράγραφος 8, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Δεύτερο τμήμα. Αρχικό κείμενο. Άρθρο 3. Παράγραφος 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Αναθεωρημένη. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 και 35. Ταυτόσιμες. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Θα προτιμούσα να κάνουμε έλεγχο δεύτερο τμήμα τροπολογία 21 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. 15. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Ονομαστική κλίση. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Ονομαστική. Πέρα. Εγκρίνεται. Πρώτη τροπολογία αναθεωρημένη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά θα προτιμούσα να ελέγξουμε. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία αναθεωρημένη υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Και τώρα η πρόταση κανονισμού όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μια καταπληκτική νομοθετική πράξη του Κοινοβουλίου. Περνάμε τώρα στο σχέδιο ψηφίσματος, στο σύνολό του, με ονομαστική ψηφοφορία. Έρχεται. Πέρας και εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Φόξ. Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για τεχνητή νοημοσύνη και την ρομποτική. Μία ψηφοφορία, ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Και εγκρίνεται. Μετά η έκθεση Γκιούτελαντ για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων 34 υπέρ κατά αποχές ε, ε απορρίπτεται παράγραφος 5 του αρχικού κειμένου μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε το μέρος δεύτερο της παραγράφου 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παραγραφός 7 του αρχικού κειμένου σε δύο μέρη υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6, μέρος πρώτο με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται μέρος δεύτερο της τροπολογίας 6, επίσης με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 σε δύο μέρη μέρος πρώτο άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται και μέρος δεύτερο της 7 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία και πέρας εγκρίνεται τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας ναι, απορρίπτεται περνάμε στο αρχικό κείμενο σε δύο μέρη παραγραφός 17 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγραφός 18, αρχικό κείμενο, άρχεται ονομαστική ψηφοφορία και πέρασε. Εγκρίνεται. 19, αρχικό κείμενο, άρχεται ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παραγραφός 20, τροπολογία 11 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται παράγραφος 22 αρχικό κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται και πέρασε εγκρίνεται μετά από την παραγραφό 24 το τοπολογία 37 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται παραγραφός 25 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 με μασική ψηφοφορία άρχεται πέρας εγκρίνεται 17 άρχεται η ψηφοφορία ονομαστική πέρας απορρίπτεται 18 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Τοπολογία 2 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται.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 Περνάμε κατόπιν στην 9. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο, τροπολογία 9, επίσης με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20D, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 48, μέρος πρώτο με ονομαστική ψηφοφορία. Μάρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο, επίσης με ονομαστική ψηφοφορία. Μάρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 21D. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε. 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 58 σε δύο μέρη. Μέρος ε, πρώτο. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο. Επίσημη ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 44 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 24 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. 61 σε δύο μέρη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Προτιμώ να το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ορίστε. Να, να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ναι, να την επαληθεύσουμε. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Έναρξη της ψηφοφορίας. Τροπολογία 28. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά εποχές ας επαληθεύσουμε την 14 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφο D, το αρχικό κείμενο τη ιδεολογικής έκθεση σε ονομαστική ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα όλο το κείμενο μαζί, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Μπέλετ. Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Άλλη μια ψηφοφορία παρακαλώ, πολύ λίγη ησυχία. Παράφος 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος μη της αιτιολικής έκθεσης υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε όλο το κείμενο στο σύνολό του ονομαστική ψηφοφορία έναρξη Πέρασε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς απόγευμα. Uh, Ξεκινούμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Παρακαλώ πολύ όποιοι θέλετε να εγκαταλείψετε την αίθουσα να το κάνετε σιωπηρά. Θα δώσω το λόγο σε τρεις συναδέλφους που έχουν ζητήσει να μιλήσουν για το θέμα της ε, Συμφωνίας Αλλιευτικής Συμπράξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της ακτής του Ελεφαντοστού. Έκθεση του συναδέλφου Ζωάου Φερέιρα. Πρώτος ομιλητής, Ίσως περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω όμως, για να εγκαταλείψουν την αίθουσα όσοι αποχωρούν. Περνάμε σε επεξηγήσει ψήφων. Καταρχήν δίνω το λόγο στα άτομα που τον ζήτησαν για το θέμα της Συμφωνίας Ελευτικής Σύμπραξης με την Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού του συναδέλφου Ζωα Ο λόγος του συνάδελφου Αγγιλέρα Γκαρσία. Ένα λεπτό. Κυρία Αγγιλέρα Γκαρσία, να διευκρινίσω για ποιο λόγο ψήφισα υπέρ. Οι συμφωνίε αλληλευτική σύμπραξη είναι πάντοτε θετικέ, πάντοτε σημαντικέ και για τι χώρε με τι οποίε θα τις υπογράφουμε, αλλά και για τον Ευρωπαϊκό Στόλο. Ειδικά όμω για αυτή τη συμφωνία, να υπογραμμίσω το εξή: πρόκειται για μια μικρή χώρα, δημοκρατία τη ακτή του Ελεφαντοστού, 20 εκατομμύρια κάτοικοι, πάνω από 60 εθνοτικέ ομάδε και μια χώρα η οποία έχει περάσει από, μια, από πολλές φουρτούνες, ε, ε πόλεμο και πολλά κοινωνικά προβλήματα. Εμφύλιο πόλεμο και κοινωνικά προβλήματα. Ο ελευτικό τομέα δεν είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη χώρα, όμω είναι πολύ θετική αυτή η συμφωνία και για τη χώρα και για μα. Επιπλέον θα ωφεληθούν ε, η, τα σκάφη μας τα οποία ψαρεύουν τόνο. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η συμφωνία και για τα δύο μέρη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αγγιλέρα Γκαρσία. Ο λόγος των συνάδελφων Χάνων. Για ένα λεπτό. Ε, τις προάλλες ήταν πάλι στην επικαιρότητα ε, με το μπέρδαμα με τις σημαίες, μετά με το με την Ιρλανδική, με το τα Ιρλανδικά σύνορα. Ε, πάση περιπτώσει, έχουμε εκατοντάδες τέτοιες συμφωνίες και επανειλημμένως έχω πει ότι όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι υπεραλλιεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα δικά μας νερά. Να δούμε και μια άλλη πτυχή και πάλι την Αφρικανική Ήπειρο τη μεταχειριζόμαστε σαν να είναι οικονομική μας απικία που θα, μας, ε, θα δίνει πρώτες ύλες στη δική μας βιομηχανία. Μπορούμε να, ε, μπορούν να εξάγουν ε, Μπορεί να εξάγουν καρπούς καφέ, αλλά όχι ψημένο καφέ οι χώρες Αφρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ και το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε θα ήταν να ε, καταργήσουμε την κοινή αγροτική πολιτική. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Σον Κέλλη. Σημαντικές ευκαιρίες ανοίγονται από αυτή τη συμφωνία για να συνεργαστούμε σε ένα με ένα βιώσιμο τρόπο στην εκμετάλλευση των αλληλευτικών αποθεμάτων. Η βιωσιμότητα είναι σημαντικό στοιχείο της αλευτικής πολιτικής. Οπότε χαίρομαι για αυτή τη συμφωνία που δίνει σημασία στη βιωσιμότητα. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της μπλε οικονομίας. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτές τις εξέλιξεις. Καλωσορίζουμε επίσης και το γεγονός ότι αυτή η συμφωνία είναι αμοιβαία ωφέλιμη. Δημιουργεί ευκαιρίες για την εκμετάλλευση αλευτικών πόρων από αλληλευτικά σκάφη που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει ότι αυτή η εκμετάλλευση θα γίνεται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Αυτό είναι προτεραιότητα. Θα προστατεύουμε το θαλάσσιο περιβάλλον και θα λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη έκθεση και πάλι του Ζωάου Φερέιρα στο, για το ίδιο θέμα. Πρόκειται για ένα ψήφισμα. Ποιο Χάνων έχει το λόγο. Α, ο κύριος Χάνων έφυγε. Οπότε περνάμε πιο κάτω. Έκθεση Σαλαφράνκα για το πρόγραμμα καταπολέμησης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρογεύσκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σντρογεύσκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είχα την ευκαιρία στην συζήτηση να αναπτύξω τις ε, απόψεις μου για το θέμα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ακριβώς είναι το σημαντικό θέμα. Πρέπει να αποφύγουμε την δημιουργία γραφειοκρατίας. Αλλά εδώ πέρα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, έτσι από αυτό το οποίο τελικά θέλαμε. Να σας ε, υπενθυμίσω πως ε, είχε μεγάλη απήχηση η έκθεση γιατί εγκρίναμε πάρα πολλές ε, τροπολογίες. Σας ευχαριστώ κύριε Στρογεύσκη. κατόπιν έχουμε τον κύριο Μαριά. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια σημαντική δράση την οποία βεβαίως πρέπει να ενισχύσουμε αυτό που έχω αναδείξει και στην ομιλία μου είναι μια ειδική μορφή απάτης που έχει σχέση με ελληνοποιήσεις αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. δηλαδή γαλακτοκομικά προϊόντα φερρυπίν γάλα εισάγεται από την αλβανία στην ελλάδα και βαφτίζεται ελληνικό. ταυτόχρονα κτηνοτροφικά προϊόντα κρέας εισάγεται στην ελλάδα από τα σκόπια και βαφτίζεται επίσης ελληνικό. αυτές οι ελληνοποιήσεις αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων είναι ειδική μορφή απάτης και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα από την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση. και εδώ χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία λείπουν και θα πρέπει να επιβληθούν ποινές στα γειτονικά αυτά κράτη και στην αλβανία και στα σκόπια στο πλαίσιο της πολιτικής της προενταξιακής που υπάρχει από πλευράς ευρωπαϊκής ένωσης. απαιτούνται μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι παράνομες ελληνοποιήσεις αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ε, ε, ε. Σας ευχαριστώ. έφυγε και μας ε, διευκόλυνε. Οπότε περνάμε στον συνάδελφο, τον κύριο Μάμικινς, που έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Η πρόσφατη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου μα δίνει του σχετικού αριθμού για το 2017 για την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 393 δισευρώ. Μόνο ένα μέρο εκατομμυρίων ευρώ, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των κονδυλίων αυτών ανακτήθηκε. Ε, πολιτικοί και οι οικογένειέ του πολλέ φορέ αποφελήθηκαν ή ε, ο τομέα τη γεωργία από κακοδιαχείριση. Ε, πλήττεται βεβαίω η αποτελεσματικότητα τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν υπάρχει πραγματικό ευρωπαϊκό μηχανισμό για την έρευνα ε, και την ανείχνευση αυτών των ποσών. Εδώ είμαστε για να καταπολεμήσουμε την απάτη. Δεν μπορούμε να επαφιόμαστε πλήρω ε, στι εθνικέ αρχέ που κάποιε φορέ είναι και αυτέ μπλεγμένε. Ε, γι' αυτό λοιπόν η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόσδεκτη. Καλωσορίζω και τι τροπολογίε στην έκθεση του κ. Σαλαφράγκα, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και σωμάτων, όπω όλα Eurojust, Ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, και γι' αυτό υπερψήφισα. Ευχαριστούμε κύριο Πόσπισιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω υπερψηφίσει την έκθεση αυτή και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που ενέκρινε τις τροπολογίες που ε, ε, βελτιώνουν την τελική εκδοχή της έκθεσης αυτής. Η καταπολέμηση της χρηματοοικονομικής απάτης που πλήττει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς Ε, είναι ε, ένα φαινόμενο που πλήττει όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα δηλαδή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν κάθε λόγο να διώξουν την απάτη στο ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι προφανώ πρέπει να υπάρξουν έρευνε ε, και μάλιστα που να φέρουν αποτέλεσμα, ώστε να υπάρχει περισσότερη χρηματοδότηση για τα σώματα και του φορεί που τη χρειάζονται. Τα χρήματα αυτά που διαφεύγουν είναι πολύ σημαντικά. Τα κονδύλια αυτά τα θέλουμε. Πρέπει όμως να έχουμε και κατάλληλα εργαλεία για να ανοιχνεύσουμε την απάτη. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω την έκθεση και ελπίζω ότι θα βοηθήσει στο σκοπό μα. Οι μελλοντικές στατιστικές ελπίζω, ελπίζω επίσης να είναι πιο χρήσιμες. Ευχαριστούμε κυρία Πόσπεσιλ. Και τώρα περνάμε στην έκθεση του κυρίου Καντέκ για το πολιετέ σχέδιο για τα αποθέματα εχθείων στα δυτικά ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα και τι ελευθερίε δραστηριότητε εκμετάλλευση των λόγων αποθεμάτων. Ο λόγο στον κύριο Μάθιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θέλω και εγώ να πω ότι με χαρά υπερψήφισα την εκθεσία αυτή που αλλάζει τον τρόπο όπου η αλληλεία ελέγχεται στα δυτικά είδατα. Νομίζω όλοι εδώ αναγνωρίζουμε ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική στην παράδοση του χρόνου έχει αποβεί καταστραφική για την ευρωπαϊκή αλληλευτική βιομηχανία. Κατέρευσαν τα αποθέματα, τα αποθέματα, προκλήθηκε ανεργία και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Τώρα λοιπόν καλό είναι να προχωρήσουμε στην μεταρρύθμιση και με μια προσέγγιση πιο περιφερειακή. Αυτή φαίνεται να είναι η μόνη λύση και καλώ αυτό προβλέπεται για τα δυτικά ύδατα και τα παρακείμενα ύδατα του, όπου βεβαίω δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα οι αλλοί τη Μεγάλη Βρετανία. Βεβαίω είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη δεν μπορεί να ε, καταφέρει να ελέγξει πλήρω την αλία ε, και μάλιστα να αναλάβει τον έλεγχο του τι γίνεται σε μικρότερους φορείς και άλλων εθνών. Εκείνοι δεν κατανοούν, ε, δεν, δεν κατανοούν την αλλήλεια, αλλά θα χάσουν πολλά αν γίνει ε, βιώσιμη. Ελπίζω ότι μετά τον Brexit θα μπορέσουμε τουλάχιστον αυτό να το πετύχουμε στην Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστούμε κύριε Μάθιους και τώρα η κυρία Αγγιλέρα Γκαρθία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχουν πολλά θετικά, αλλά το πιο θετικό είναι ότι υιοθετήθηκε πριν το Brexit ε, αυτό το σχέδιο. Οπότε τα δυτικά ύδατα του Ατλαντικού θα ρυθμιστούν με ένα πολιετές ε, σχέδιο ε, για τα αποθέματα και καταφέραμε και τον κρίναμε πριν γίνει το Brexit. Θετικό αυτό λοιπόν διότι θα δώσει καλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στον ελευτικό τομέα. Καταρχήν θα θέλαμε να είχε γίνει διάκριση ανάμεσα στο βορρά και το νότο, αλλά ακόμα και έτσι τελικά ε, θα εξασφαλίσει αυτή τη σταθερότητα στον ελευτικό τομέα. Μιλάμε για παραπάνω από 4.000 αλληλευτικά σκάφη σε ένα πολύ σημαντικό λοιπόν κομμάτι του κόσμου. Θα θέλαμε να είχε περιοριστεί περισσότερο η εραστεχνική αλία έναντι της ε, επαγγελματικής αλίας, αλλά σε κάθε περίπτωση Το σχέδιο αυτό, το πολιετές αυτό σχέδιο είναι πολύ θετικό για το μέλλον της αλίας στον Ατλαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγγιλέρα Γκαρσία. Ο λόγος του Σον Κέλλη. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι μόνο η Αλία στα δυτικά ύδατα, γιατί έχουμε μια πολύ καλή συμβαστική πρόταση στα χέρια μα. Θα βοηθηθούν οι Αλίες μα που δραστηριοποιούνται στι θάλασσε να συνεχίσουν τη δραστηριότητά του αλλά με τρόπο που θα επιτρέψει να προστατευτούν και τα αποθέματα και το περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν μπορούμε να ψαρέψουμε όλα τα ψάρια. Αυτό είναι η ουσία. Μετά δεν θα έχουμε κανένα ψάρι για το μέλλον και δεν θα έχουμε και ψαράδες. Άρα η συμβαστική πρόταση είναι η καλύτερη λύση και την καλωσορίζω. Επίσης, καλωσορίζω τη συμφωνία για την ε, ψυχαγωγική αλία και αυτό είναι σημαντικό και το ψήφισμα αυτό, θα, η έκθεση αυτή θα βοηθήσει και τους ανθρώπους αυτούς στο σκοπό τους, καθώς και την ε, διάσταση του τουρισμού. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερος προσωπικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη ε, και τώρα να περάσουμε στην επόμενη έκθεση. Έκθεση της συναδέλφου Γκαρντίνη για τον μηχανισμό προλητικής προστασίας της Ένωσης. Δύο συναδέλφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μάουλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ μια πτυχή που έχει οδηγήσει σε σύγχυση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης διαθεσιμότητα ε, Ιδίω ω προ την οικονομική βοήθεια προ το μηχανισμό πολιτική προστασία. Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα λεπτή, ιδίω από την άποψη τη απασχόληση, γιατί είναι δεκάδε τα εκατομμύρια άνεργοι σε όλη την Ευρώπη, ε, ιδίω στι χώρε τη Μεσογείου και την Ιταλία όλο ιδιαίτερω. Η ε, η κατάσταση είναι πια ένα κοινωνικό ε, καθεστώ Έχει θεσμοθετηθεί. Το Κοινοβούλιο λοιπόν σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη στιγμή που περνάει η Ευρώπη θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτούς που εκπροσωπούν τα θεμέλια της ενώσης μας, την εθνική μας ταυτότητα. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω όλα αυτά να οδεύσουν προς τη σωστή κατεύθυνση και όχι απλώς την σωστή, και να μην ασχοληθούμε μόνο με την υπέρμετρη, κάποιε φορέ υπερβολική προστασία των μειονοτήτων ε, που βρίσκονται στην υπερό μα. Εντάξει, έχουν και αυτοί δικαιώματα, πρέπει να ενταχθούν, όμω ε, δεν έχουν τη διάθεση ούτε να βοηθήσουν να κάνουμε όσα του ζητούμε, δηλαδή να συνεργαστούν. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μαριάς τώρα. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια σημαντική δραστηριότητα διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω οι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα λόγω φυσικών καταστροφών. Στην Ελλάδα είχαμε τις ε, φωνικές ε, πλημμύρες στη Μάντρα της Αττικής, είχαμε τις φωνικές ε, πυρκαγιές ε, στο μάτι πάνω από 100 νεκροί και ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει οι πληγέντες τις αποζημιώσεις τους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, να ενσκύψει η κυβέρνηση η οποία λόγω της ανικανότητας που την διακρίνει δεν έχει ακόμη χορηγήσει τις αποζημιώσεις στους ίδιους τους πληγέντες φυσικά θα πρέπει να προβλέψουμε και αλλαγές στην διαδικασία της λειτουργίας του περίφημου ταμείου αλληλεγγύης διότι οι προϋποθέσεις πρέπει να γίνουν πολύ πιο ευέλικτες για να υπάρχει η δυνατότητα της ε, καταβολής των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε κάποιον ακόμα που έχει ζητήσει το λόγο. Συνάδελφο ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν περισσότερε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τον συντονισμό των δυνατοτήτων απόκριση, ε, πολιτική ε, προστασία και ανθρωπιστική ε, αντίδραση από το όσα προέκυψαν τα τελευταία χρόνια που μα τα δείχνουν ξεκάθαρα. Πρέπει να δημιουργηθεί αυτό ο μηχανισμό που ήδη έχει λειτουργήσει στην Πορτογαλία. Βρισκόμαστε σε μια φάση διαπραγματεύσεων για να δούμε πόσο εμπορικά μπορεί να τεθεί η οργάνωσή του και να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρω για να αντιμετωπίσει τι ανάγκε συνεργασία μεταξύ μελών. Γι' αυτό λοιπόν έχει φτάσει η στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι ένα Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτική Προστασία μπορεί να προωθήσει μια συλλογική απάντηση τη Ευρώπη πιο ισχυρή, αναλαμβάνοντα ένα συγκεκριμένο και αποφασιστικό ρόλο για τον σχεδιασμό μια κοινή στρατηγική που μπορεί και σε καιρού ειρήνη να δώσει γρήγορη απόκριση στι συνέπειε των κλιματικών αλλαγών, στι ανθρωπιστικέ ανάγκε και όσα έχουμε δει να προκύπτουν στι τελευταίε ημέρε. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό ε, υπάρχει ανάγκη να κάνουμε καλύτερο και ε, πιο ισχυρό ε, το ε, του rescue, ώστε, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση, την έκθεση Μποναφέ για τις ελάχιστες απαιτήσει ε, για την επαναξυποποίηση των υδάτων. Ο κύριος Σόλτες πρώτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να είμαστε σαφείς, οι υδάτινοι πόροι υφίστανται πίεση, γι' αυτό είναι το σημαντικό αυτό το οποίο κάναμε εδώ πέρα σήμερα. Το... Η ύδατα είναι μεγάλη πρόκληση και θα είναι μεγάλη πρόκληση στο μέλλον, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων. Βεβαίω, η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων απαιτεί υποδομές ε, εγκαταστάσει βιολογικού καθαρισμού και βεβαίω ε, θα επηρεάσει την γεωργία. Θα μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τα ύδατα στην γεωργία και υπάρχουν και κάποιες νέες καλλιέργειες. Πρέπει λοιπόν να επαναξιμοποιηθεί αυτό το νερό για γεωργικούς σκοπούς. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος ο κύριος Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήμουν πρόεδρος, δήμαρχος του Πρότσλαβ, οπότε ξέρω το πρόβλημα. Και το αναφέρω αυτό γιατί η έκθεση αυτή ε, πραγματικά εισάγει μια σημαντική καινοτομία. Ο εισηγητής χρησιμοποιεί, συμφωνεί με τη χρήση κυρίως στην Γεωργία, όμως πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση και στην επαναξιμοποίηση των αστικών υδάτων. Το αναφέρω